Καλημέρα σας. Αρχίζει η, ε, η Ολομέλεια, η ημερήσια διάταξη προβλέπει την έκθεση της κυρίας Νικόλ Κιλ Νίλσον για τις γυναίκες και την κλιματική αλλαγή. Έχετε τέσσερα λεπτά, κυρία Συγήτρια. Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και εκφράζω την ικανοποίησή μου για όλες τις ε, πολύ ενδιαφέρουσες συνεισφορές ε, σε αυτήν την έκθεση. Ελπίζω ότι έτσι θα μπορέσουν να συνειδητοποιήσουν τα προβλήματα τα θεσμικά όργανα. Σε ένα ιδανικό κοινοβούλιο δεν θα υπήρχε μια επιτροπή γυναικών, διότι εγκαρσίως όλα τα γυναικεία προβλήματα και προβληματικές θα επισύρχονται σε όλες τις άλλες πολιτικές. Αλλά εδώ χρειάζεται κάθε φορά να παλεύουμε για να πείσουμε τους συναδέλφους, γιατί εμείς της Επιτροπής Γυναικών θέλουμε να βγάλουμε τις γυναίκες από το σκούρο σημείο των πολιτικό, κοινοτικών πολιτικών και για τα περιβαλλοντικά θέματα. Εμείς στην έκθεσή μας θέλουμε να αποδείξουμε ότι οι γυναίκες ε, δεν είναι τα πράσινα φυτά της ε, οικολογίας. Οι γυναίκες ε, κινδυνεύουν 14 φορές περισσότερο να πεθάνουν σε θεομηνίες, πόσο μάλλον στο τσουνάμι ή στην, ε, στον καύσωνα στην Ευρώπη, όπου το μεγαλύτερο ποσοστό θυμάτων ήταν οι γυναίκες. Και αυτό γιατί οι γυναίκες δεν έχουν τα ίδια οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά μέτρα να προσαρμοστούν ή να διαφύγουν. Στην, Ονδου, στην Ονδούρας η πόλη της Λαμασίκα που κατάφερε να προστατεύσει τις γυναίκες με συγκεκριμένα μέτρα δεν είχε κανένα θύμα όταν ε, ήρθε ένας κυκλώνας. Βλέπουμε όμως ότι δεν είναι μόνο η οικολογία η οποία υποφέρει, τα δικαιώματα των γυναικών είναι αυτά που υποφέρουν παράλληλα. Γι' αυτό συνδυάζοντας τα δύο εμείς θέλουμε να προτείνουμε αποτελεσματικά μέτρα σε κάθε κρίση ή σε κάθε ε, σύραξη λέγανε τα, ανθρώπινα, τα γυναικεία δικαιώματα έρχονται μετά. Κάθε φορά έρχονται μετά. Τα οικολογικά προβλήματα όμως με τα προβλήματα των γυναικών συνδέονται άμεσα. Δεν είναι όμως μόνο θύματα που πρέπει να προστατεύσουμε οι γυναίκες. Έχουν και προτάσεις να υποβάλουν. Διότι αυτό όμως δεν συμβαίνει διότι ζούμε σε καθαρά φιλετικές κοινωνίες. Το να είναι κανείς άντρας ή γυναίκα έχει επιπτώσει στην καθημερινή μας ζωή για την ε, επιλογή ε, του επαγγέλματος, ε, για την πρόσβαση στους πόρους, για τις ιδέες που μπορεί να προτείνει. Εμείς έχουμε προβλέψει τέσσερα μέτρα εκπροσώπησης. Πρώτον, Ζητούμε 40% γυναίκες σε πολιτικές, οικονομικές και τεχνικές αρχές. Η φωνή των γυναικών πρέπει να υποστηρίξει. Δεύτερο, προστασία και κατάρτιση. Να έχουμε έναν ειδικό κύκλο για τις γυναίκες όπου από θύματα γίνονται πρωταγωνιστές των αλλαγών. Για κατάρτιση, για να ξεκινήσει η οικονομική η πράσινη οικονομία για να μπορέσουν οι γυναίκες να προχωρήσουν στην τεχνολογική προσαρμογή και στις αλλαγές που είναι απαραίτητες και μετά έρευνα χρειαζόμαστε στοιχεία αναφύλλω για να βελτιώσουμε την κατανόηση του θέματος και τις πολιτικές μας προτάσεις. Για να ολοκληρώνω στο πνεύμα αυτής της έκθεσης, λέω ότι η πολιτική καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών θα πρέπει να εμπλουτιστεί εντάσσοντας το ζήτημα των φύλων και καταπολεμώντας τις διακρίσεις για να έχουμε και θα έχουμε έτσι και αποτελεσματικότερες πολιτικές για το περιβάλλον. Μπορούμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε με, αυτόν τον τρόπο ένα μια τέτοια σημαντική πρόκληση όπως είναι οι κλιματικές αλλαγές. Φτάνει να έχουμε και τους πόρους για να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ Εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Ποτότσνικ, για τρία λεπτά. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εξ ονόματος της Κομισιόν και ιδιαίτερα του συναδέλφου μου Κόνι Χέρεγκαρτ που δυστυχώς δεν μπορεί να παρίσταται σήμερα, χαιρετίζω την έκθεση για τις γυναίκες και την κλιματική αλλαγή και ευχαριστώ την εισηγήτρια για την εξαιρετική της εργασία καθώς και για όλα μας όσα μας είπε. Είναι πολύ καλή αυτή η ευκαιρία συζήτησης του πώς θα μπορούσε η Ένωση να βοηθήσει τις γυναίκες γιατί οι κλιματικές αλλαγές είναι γεγονός για πολλούς κατοίκους του πλανήτου, ιδιαίτερα στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Όπως γνωρίζετε, περισσότερο πλήττονται οι πτωχότεροι και οι πιο αδύναμες κατηγορίες του πληθυσμού μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά όπως λέει σωστά και η έκθεση, δεν αφορά συγκεκριμένα φύλλα η κλιματική αλλαγή, αλλά πλήττει διαφορετικά. Θα πλήττει διαφορετικά. Παραδείγματο χάρη, <clears throat> ο τρόπος ζωής και κατανάλωσης είναι διαφορετικός. Αν τονίσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη με χαμηλές εκπομπές διοξιδίου, ενισχύουμε ολόκληρη την οικονομία και βοηθάμε έτσι και τους ασθενέστερους όπως τις γυναίκες και τους παιδες με τα γεωγραφικά και θεματικά μας προγράμματα θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε παραδείγματο χάρη αυτή τη Σαββατοκύριακο οργανώνεται στις Βρυξέλλες η διάσκεψη για την ε, βιώσιμη ενέργεια για όλους μεταξύ των θεμάτων είναι και η καλύτερη χρήση της βιομάζας για το μαγείρεμα. Επίσης θα αφήσει περισσότερο ελεύθερο χρόνο για τις γυναίκες που δεν θα χρειάζεται τόσο πολύ για να συλλέγουν προσανάματα ας πούμε. Επίσης στοχεύει η Ένωση να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της πρόβλεψης θεομηνιών και άλλων κινδύνων που μπορεί να επηρεάζουν τα φύλλα στις συνέπειές τους. Η ισότητα των φύλων και η ισότιμη μεταχείρισή τους είναι από τους βασικότερους στόχους που έχουν εγκριθεί από την Ένωση γενικά. Και όπως λέει και η έκθεση, τα προγράμματα που δεν λαμβάνουν υπόψη τα φύλλα πρέπει καταρχήν να διασφαλίζουν την ισότητα από άλλα μέσα για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για ουδετερότητα. Οι γυναίκες είναι η πλειοψηφία των πτωχοτέρων κατοίκων του πλανήτη αλλά υποεκπροσωπούνται παντού και στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Κατά τη συζήτηση της νέας εταιρική σχέσης Ένωσης Ειρηνικού είχαμε πει ρητά ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν οι κλιματικές αλλαγές στην περιοχή εκείνη ιδίως του Ειρηνικού όπου υπάρχει ιδιαίτερη υποεκπροσώπηση των γυναικών. Οι ηγέτες των χωρών του Ειρηνικού αναγνωρίζουν ότι οι γυναίκες γνωρίζουν καλύτερα τα πράγματα στις πρακτικές λεπτομέρειες της ζωής για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άρα και για τη δημιουργία οικονομικής ανάπτυξης. Σε συμφωνία λοιπόν με τον στόχο 40% εκπροσώπησης των γυναικών τέθηκε το θέμα της ισότητας των φύλων και στις τελευταίες διασκέψεις του οηές ή FCCC που λέμε. Πρέπει λοιπόν η Ένωση να διασφαλίσει όσο το δυνατόν καλύτερα την ισότητα των φύλων. Η Δανική Προεδρία μας ανέφερε ορισμένους δείκτες που σκοπεύει να καταθέσει στο Συμβούλιο μεταξύ των οποίων και ο δείκτης για την ισότητα των φύλων που είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε και να αποτιμήσουμε τα πράγματα. Θα χρειαστεί χρηματοδότηση, capacity building και έτσι θα μπορέσουν οι γυναίκες να βελτιώσουν τη ζωή τους διότι η δική μας ευθύνη είναι να τους δώσουμε μια θέση και για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Η σημερινή λοιπόν έκθεση είναι πολύ χρήσιμη και ελπίζω να εγκριθεί. Ε, συγχαίρω δε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρωτοβουλία του και καταλήγω με τα εξή θετικά. Πιστεύω ότι η αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών μπορεί να βελτιώσει τα πράγματα και τις συνθήκες διαβίωσης ανδρών και γυναικών στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Η Κομισιόν θα συνεχίσει να προσέχει τα θέματα της ισότητας των φύλων και στο θέμα της καταπολέμησης των κλιματολογικών αλλαγών. Σας ευχαριστώ. Και τώρα, εξ ονόματος της Επιτροπής Περίβ, θα ακούσουμε την κυρία Λιωτάρα. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια. Οι φτωχότεροι του πλανήτη είναι κατά 70% γυναίκες και όπως είπε ε, ο Επίτροπος και η εισηγήτρια αυτές χτυπάει η κλιματική αλλαγή. Ε, είναι τα μεγαλύτερα θύματα σε φυσικές καταστροφές αλλά και σε πολέμους. Περιέργως δε και κατά τρόπο ηρωνικό βρίσκονται λίγες γυναίκες στα κέντρα αποφάσεων για την κλιματική αλλαγή, γιατί δεν, είναι, ε, δεν εκπροσωπούνται μεταξύ των εμπειρογνωμόνων. Θεωρώ πως μπορούν να προσφέρουν πολλά σε μια καλύτερη κλιματική πολιτική. Δεν υπάρχει ακόμα γνώση για την ισότητα των φύλων στο κλίμα, αλλά σίγουρο είναι πως ε, είναι καλύτερη για το κλίμα η μεγαλύτερη ισότητα και συνεισφέρει και το καλύτερο κλίμα στην ισότητα. Και σκεφτούμε το ότι δεν θα πηγε, πρέπει να πηγαίνω έρχονται να κουβαλάνε νερό και ξύλα όπως είπε ο Επίτροπος και δεν θα μπορούν έτσι ε, να μαθαίνουν να διαβάζουν. Γιατί μην ξεχνάτε πως ένα έξυπνο κορίτσι που έχει πάει σχολείο είναι προετοιμασμένο για την κλιματική αλλαγή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξ ονόματος ε, των ομάδων, η κυρία Νεδέλτσεβα για το ΕΛΚ. Εγώ θα ήθελα αγαπητοί συνάδελφοι να συγχαρώ την κυρία Κιλ Νίλσεν ε, για τη δουλειά της όπως επίσης και τους κοιόδης εισηγητές ε, για την συνεισφορά τους σε αυτή την έκθεση για την προστασία ε, για τις γυναίκες συγγνώμη, και κλιματική αλλαγή. Πάνω από το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού αποκλείεται από τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες πλήττονται άμεσα από τις επιπτώσεις των περιβαλλοντικών πολιτικών και είναι αυτές που γνωρίζουν καλή, τις ε, βέλτιστες πρακτικές καλύτερα από όλου. Θα πρέπει λοιπόν οι γυναίκες να είναι πρωταγωνιστές ε, των αλλαγών για την προστασία του περιβάλλοντος. Πιστεύω ότι η προστασία του περιβάλλοντος περνάει και από τη συμμετοχή των γυναικών στην μελέτη όλων αυτών των προβληματικών. Θα πρέπει να ανοίξουν οι επιστημονικοί κλάδοι για τις γυναίκες αυτούς τους τομείς θα πρέπει να προωθήσουμε τις ε, γυναίκες ε, στα κέντρα λήψης αποφάσεων για να μπορούμε να λαμβάνουμε μεγαλύτερες, περισσότερες πράσινες λύσεις για τη διαχείριση των, περιβαλλοντικών προβλημάτων. Η ισότητα των φύλων και από περιθωριοποίηση των γυναικών στο πλαίσιο της αηφορίας συμμετοχή των γυναικών στην διαχείριση των περιβαλλοντικών προβλημάτων ε, με τις γυναίκες πρωταγωνιστές στην προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό θα επιτρέψει στις γυναίκες να έχουν και μεγαλύτερη πρόσβαση στους οικονομικούς και φυσικούς πόρους. Κερδίζουν όλοι από αυτές τις πολιτικές Χρειάζεται ένα σύνδεσμος μεταξύ προστασίας της, του περιβάλλοντος και ισότητας των γυναικών. Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος των σοσιαλιστών η κυρία Εστρέλα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ θα ξεκινήσω συγχαίροντας την κυρία Κιλ Νίλσεν η οποία συνέταξε μια πολύ ενδιαφέρουσα και καλώς διαρθρωμένη έκθεση. Η καλή συνεργασία με τους σκιώδης εισηγητές οδήγησε σε μεγάλη συνένεση. Οι κλιματικές αλλαγές δεν είναι ουδέτερες όσον αφορά στα φύλλα, διότι δεν πλήττουν κατά τον ίδιο τρόπο άντρες και γυναίκες φτωχούς ή πλούσιους, αναπτυγμένες ή αναπτυσσόμενες χώρες. Η κλιματική αλλαγή φαίνεται πολύ περισσότερο στις πιο φτωχές χώρες, εκεί όπου οι κοινωνικές ανισότητες είναι μεγαλύτερες και οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια. Το 70% των φτωχών είναι γυναίκες και κατά συνέπεια είναι και οι πιο ευπαθείς στις κλιματικές αλλαγές και στις θεομηνίες ο αγώνας κατά της κλιματικής αλλαγής συνδέεται άμεσα με την ισότητα των φύλων. Οι θεομηνίες έχουν άμεσες επιπτώσεις μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα στα ζητήματα που αφορούν στην εκπαίδευση, στην μετακίνηση των πληθυσμών και οι νέες γυναίκες είναι ιδιαίτερα ευπαθείς εναντί των θεομηνιών όπου έχουμε μεγαλύτερες θεομηνίες η συμμετοχή η, η εκπαίδευση των γυναικών είναι πολύ μικρότερη η, η ξηρασία, η έλλειψη νερού υποχρεώνουν τις γυναίκες να εργάζονται περισσότερο για να εγγυθούν το νερό, την διατροφή και τα κορίτσια, τα νέα κορίτσια εγκαταλείπουν το σχολείο για να βοηθήσουν τις μαμάδες τους που ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Χρειάζονται λοιπόν μέτρα τα οποία να ενσωματώνουν την διάσταση των φύλων στην στρατηγική πρόβλεψη των θεομηνιών. Οι γυναίκες είναι συνηθισμένες να διαχειρίζονται τους φυσικούς πόρους. Δεν πρέπει εμείς να αγνοούμε αυτή τη δυναμική για την βελτίωση των στρατηγικών για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Ο κύριος Γιώχανσον. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για το έργο της. Είναι πολύ σημαντική αυτή η έκθεση και η δική μου συνεισφορά αφορά ακριβώς τα θέματα αυτά και την συνένεση εντός, και τη συνένεση εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των λοιπόν Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων για τα θέματα αυτά. Οι γυναίκες έχουν λιγότερη πρόσβαση στους πόρους, την εκπαίδευση και ε, οι γυναίκες και τα παιδιά πλήττονται σκληρότερα από την κλιματική αλλαγή. Τρία τέταρτα των προσφύγων παγκοσμίω είναι γυναικόπαιδα και για να βελτιωθεί η κατάσταση χρειαζόμαστε μέτρα μεγάλης και μικρής κλίμακας. Χωρίς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση θα χάσουμε καλές ιδέες. Οι γυναίκες καταναλώνουν με πιο αηφόρο τρόπο και είναι πιο φιλικές προς το κλίμα από τους άντρες και θα αναπτύξουν νέους έξυπνους τρόπους χρήσης ε, του νερού και της ενέργειας. Χρειαζόμαστε υπεύθυνη χρήση των πόρων σε κάθε σπίτι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι στην πρωτοπορία της χρήσης των ιδεών των γυναικών και των πόρων για να μπορέσουμε να εστιάσουμε ε, στις ε, κλιματικές προκλήσεις. Ακριβώς οι γυναίκες αν συνεργαστούν θα μπορέσουν να εγγυηθούν ε, δίκαιη στρατηγική στον τομέα αυτών. Παραδείγματο χάρη χρειάζεται καλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών στους φορείς ε, λήψης αποφάσεων π.χ. στις σχετικές διαπραγματεύσεις. Σας ευχαριστώ για τους Ευρωπαίους συντηρητικούς. Ε, τώρα η κυρία Γιανακουδάκη. επιτεύχθηκε στην τελευταία διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή χάρη σε μια συμφωνία χάρη σε δύο γυναίκες. Την ε, Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ε, Υπουργό Περιβάλλοντος της Ινδίας. Επικεφαλής ήταν επίσης η Υπουργός Εξωτερικών της Νοτιοαφρικής. Όμως η έκθεση αγνοεί τα επιτεύγματα αυτών των γυναικών. Η έκθεση αυτή μειώνει την επιτυχία του σε ένα νούμερο και ζητάει 40% ποσόστοση για γυναίκες στις διαπραγματεύσεις. Έχω εξηγήσει εδώ πολλές φορές πως οι ποσοστώσεις πατρονάρουν τις γυναίκες. Όμως εξακολουθεί να υφίσταται αυτή η παράνοια των ποσοστώσεων στην πολιτική και στις επιχειρήσεις. Και τώρα για τους εραστές των ποσοστώσεων πάμε και στις κλιματικές διαπραγματεύσεις οι ποσοστώσεις μειώνουν τις γυναίκες που τα κατάφεραν να φτάσουν στην κορφή γιατί ήταν απλά οι καταλληλότερες. Η κλιματική αλλαγή είναι μια παγκόσμια πρόκληση και χρειαζόμαστε παγκόσμιες συμφωνίες. Σας ευχαριστώ. Τώρα για την Ευρώπη, της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας, ο κύριος Χέλμερ για ένα μισή λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, εδώ πρόκειται για μια ηρωική προσπάθεια να σεβαστούμε ε, από τις κύριες μανίες του κοινοβουλίου μας. Να συνδέσουμε δηλαδή την κλιματική αλλαγή με τις γυναίκες. Αλλά δυστυχώς πρόκειται για αποτυχία. Δεν πιστεύουν και πολλοί ότι η οικιακή βία κατά των γυναικών οφείλεται ή προκύπτει από την ε, κλιματική αλλαγή και τέτοια πράγματα. Γιατί δεν κάνουμε και μια έκθεση για τους άντρες και την κλιματική αλλαγή αφού ζουν μαζί με τις γυναίκες και υφίστανται τα ίδια προβλήματα. Χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο ηλεκτρονικά μηχανήματα, τηλεόραση, υπολογιστές και εκπέμπουν διοξίδιο του άνθρακος. Η έκθεση όμως κάνει και μία σωστή διαπίστωση ότι οι γυναίκες δεν αντιμετωπίζουν σωστά όλα αυτά τα προβλήματα η μεγαλύτερη επίπτωση της θέρμανσης του πλανήτη είναι πόσο ζημιώνουν τα δικά μας προγράμματα μείωσης των εκπομπών των πλανήτη και την απασχόληση, πράγμα το οποίο καταλήγει σε μετεγκαταστάσεις σε χώρες που έχουν ακόμη χαμηλότερα κριτήρια προστασίας του περιβάλλοντος. Και δυστυχώς αυτό τελικά καταλήγει να πλήττει περισσότερο και τις γυναίκες και Το καλύτερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε για τις γυναίκες και τους φτωχούς, καθώς και για όλη την ανθρωπότητα, θα ήταν να καταργήσουμε όλες αυτές τις παρανοϊκές κλιματολογικές πολιτικές. Ευχαριστούμε. Και τώρα για την ΚΟΕ ο κύριος Γούσταυσον για δύο λεπτά. Πρόεδρε, καταρχάς ευχαριστώ την κυρία Νίλσον για την εξαιρετική της εργασία και για τη συνεργασία μας, διότι η έκθεση αυτή έχει ιστορική σημασία. Είναι η πρώτη φορά που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζει θέματα κλιματικά από την άποψη των φύλων διότι δεν έχει τις ίδιες επιπτώσεις επί των φύλων. Μπορεί να συμβάλλουν περισσότερο οι άντρες στο πρόβλημα, αλλά οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο. Ο τρόπος ζωής ευθύνεται γι' αυτό. Οι γυναίκες καταναλώνουν με πιο βιώσιμο τρόπο και επίσης είναι πιο πρόθυμες να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό του περιβάλλοντος οι σημερινές αδικίες θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο αν δεν αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των κλιματικών αλλαγών που θα πλήξουν τις φτωχότερες χώρες και ιδιαίτερα τις γυναίκες αυτές. Επομένως, η άνηση μεταχείριση υπέρ των ανδρών που ισχύει παντού ισχύει και για τις συζητήσεις στο, για τις κλιματολογικές αλλαγές και γι' αυτό ζητάμε ποσοστώσεις και στοχευμένα μέτρα για να αυξηθεί η εκπροσώπηση των γυναικών. Η Ένωση πρέπει να πρωτοπορήσει με το καλό παράδειγμα εδώ. Είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες οι γυναίκες για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και πολλά παραδείγματα δείχνουν ότι η σωστή εκπαίδευση των γυναικών μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο να μειώσει την απερίμωση και την αποδάσωση και την αποψήλωση των δασών. Όποτε ενδυναμώνονται οι γυναίκες ενδυναμώνεται ολόκληρη κοινωνία και αυξάνεται η δημοκρατία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. τον, δεν βλέπω τον κύριο Νίκ Γκρίφιν, γι' αυτό θα δώσω το λόγο. Θα δώσω λέγω τον λόγο, αλλάζοντας το... Α, ήρθε ο κύριος Γκρίφιν. Πρώτα όμως θα μιλήσει η κυρία Γιωχάνας Πιοσλεύκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όταν μιλάμε για τις γυναίκες και την κλιματική αλλαγή, είναι κάτι το καινοτόμο. Λαμβάνουμε υπόψη το γεγονός πως οι γυναίκες ε, είναι πάρα πολύ σημαντικές όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για τα εσωτερικά ζητήματα και βεβαίως είναι πιο δραστήριες στην κοινωνία των πολιτών. Θεωρώ πως πρέπει να δώσουμε περισσότερη προσοχή σε αυτό το φαινόμενο. Εάν σκεφτούμε το πώς μπορούν οι γυναίκες να εμπλακούν περισσότερο στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής, θεωρώ πως μπορεί να γίνει το εξής. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός εξή. που ε, εκπαιδεύονται ειδικά σε πολυτεχνία. Έτσι θα μπορέσουν να γίνουν ειδικοί και να απασχοληθούν σε τομείς που εμπλέκονται άμεσα με την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Επίσης, ε, Μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός των γυναικών που λαμβάνουν αποφάσεις. Η πολιτική στρατηγική πρέπει να λάβει υπόψη την ε, θέση των γυναικών, ειδικά όταν μιλάμε για ίση πρόσβαση στην ε, λεγόμενη αυτή οικονομία. Πέρα δε από τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές χρειαζόμαστε καθημερινές αλλαγές που θα αυξήσουν τη δυνατότητα των γυναικών όταν μιλάμε για την πρόσβαση σε μικροπιστώσεις. Ε, θεωρώ λοιπόν πως οι γυναίκες με πρόσβαση σε μικροπιστώσεις και τις σχετικές υπηρεσίες ε, μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο σε μια οικοοικονομία για τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο επόμενος ε, είναι η κυρία Νταντσίλα για να μισή λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα είναι η κλιματική αλλαγή και αυτό συνδέεται άμεσα με την ισότητα των φύλων. Εμείς θα πρέπει να προσπαθήσουμε ώστε οι γυναίκες να μην πεθαίνουν 14 φορές παραπάνω από ότι οι άντρες πράγμα το οποίο μας αποδεικνύουν σήμερα οι στατιστικές. Οι γυναίκες είναι οι φτωχότερες στον κόσμο, κατά 70% είναι αγρότησες και το 80% των θυμάτων είναι γυναίκες. Το μεγαλύτερο ποσοστό των προσφύγων για περιβαλλοντικούς λόγους είναι οι γυναίκες. Είναι τα θύματα της βίας που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή υπόκεινται διακρίσεις στην πρόσβαση των πόρων και στις τεχνολογίες, σε όλες τις υπηρεσίες, για τα φάρμακα. Δεν είναι ιδιοκτήτριες των χωραφιών τους, δεν μπορούν να έχουν επιστώσεις. Δύσκολα λοιπόν μπορούν να προσαρμοστούν λόγω αυτών των συνθήκων στις κλιματικές αλλαγές. Εμείς θα πρέπει να μην εντείνουμε τον ανταγωνισμό μεταξύ ανδρών και γυναικών αλλά να βρούμε τις καλύτερες λύσεις ούτως ώστε να προχωρήσουμε με τον καλύτερο τρόπο σε αυτό το πεδίο. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια τράπεζα δεδομένων αναφύλω για να μπορέσουμε να αξιολογούμε πριν ξεκινούμε τα σχέδια. Πρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα τη διάσταση των φύλων στην κλιματική αλλαγή για να βρούμε και τις καλύτερες λύσεις για να την καταπολεμήσουμε. Ευχαριστώ. Κυρία Παραμπάνοβα για ένα μισή λεπτό. Κύριε Επίτροπε, κυρίε και κύριοι, θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Νίλσεν για την εξαιρετική δουλειά τη και χαιρετίζω την έκθεση αυτή που ζητάει και μεγαλύτερο ρόλο των γυναικών για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, γιατί πιστεύω ότι το θέμα τη ισότητα των φύλων και για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος θα ήταν κάτι αποτελεσματικότερο διότι οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο από τις κλιματικές αλλαγές και από τις θεομηνίες ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το θέμα αυτό μέσα στην ευρωπαϊκή πολιτική αντιμετώπιση των κλιματικών ελλαγών και των μέτρων καταπολέμησης θεομηνιών να βασίζονται όλα αυτά και σε φιλετική στόχευση. Να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο τις δυνατότητες των γυναικών και να εφαρμόσουμε στοχευμένες προγράμματα αντιμετώπισης. Αναγνωρίζουμε βέβαια τη σημασία που έχει η διαφορετική μεταχείριση των φύλων, αλλά πρέπει να βάλουμε δεσμευτικές ρήτρε διεθνώς. Πρέπει η Ένωση λοιπόν να λύσει, να έχει προτάσεις για την παγκόσμια αντιμετώπιση του προβλήματος, α και σε δεύτερη φάση να ζητήσει μία δεσμευτική συμφωνία ή συνθήκη που να, συμπεριλα... που να περιλαμβάνει και το θέμα της διαφορετικής στόχευσης για τα φύλλα. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα ο κύριος Γρίφιν. Κύριε Πρόεδρε, είναι εύκολο να χλεβάσει κανείς αυτή την έκθεση. Μάλιστα γελάνε εκατομμύρια Βρετανοί αναγνώστες εφημερίδων. Τη στιγμή που η καταστροφή του ευρώ οδηγεί τον κόσμο στην αυτοκτονία, έχουμε εδώ πέρα συνθήματα πολιτικής ορθότητας και θα μπορούσε κανείς να το περάσει για πρωταπερλιάτικο αστείο. Αλλά στην πραγματικότητα η προσπάθεια αυτή να θεσμοποιηθεί η διάκριση εις βάρος του μισού πληθυσμού της Ευρώπης δεν είναι καθόλου αστείο. Συγχαίρουν οι γυναίκες η μία την άλλη η πρόταση αυτή είναι μια προσπάθεια να υπάρξει διχόνοια μεταξύ των δύο φίλων να καταστραφούν οι αρχές της οικογένειας και να εξαγάγουμε τις ε, αξίες αυτές παγκοσμίω. Η προσπάθεια αυτή να ε, διασπείρουμε το μίσος δεν είναι χωρίς θύματα. Εκατοντάδες χιλιάδες άντρες δεν ε, έχουν πρόσβαση στα παιδιά τους μετά τα, διαζύ... μετά τα διαζύγια χιλιάδες παιδιά αρπάζονται από το κράτος και τις οικογένειές τους ε, χάρη στον μαχητικό φεμινισμό. Εν τω μεταξύ υπάρχουν στον πραγματικό κόσμο πραγματικά προβλήματα και οι ψηφοφόροι αναμένουν να τα λύσουμε. Όχι να σπαταλάμε τα λεφτά τους σε μπουρδες σεξιστικές κατά των ανδρών. Ας σταματήσουμε λοιπόν αυτά τα κενά συνθήματα και συνεργαστούμε σε κάνα πραγματικό πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής ε, Στρίφλερ για δύο λεπτά. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Αυτή η θεματική θα πρέπει να εξεταστεί όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο και είναι αλήθεια ότι οι γυναίκες είναι τα πρώτα θύματα των κλιματικών αλλαγών η συνεχής διάκριση των γυναικών σε επίπεδο εισοδήματος, πρόσβαση των πόρων σε πολιτικό επίπεδο είναι μερικοί από τους παράγοντες που εξηγούν την ευπάθεια των γυναικών κατά την φάση των ε, θεομηνιών. Οι κλιματικές πολιτικές δεν μπορούν να γνωρίσουν τους τους ανθρώπους ε, δεν μπορούν να αγνοήσουν τα σχέδια, τα αναπτυξιακά σχέδια, το ρόλο των γυναικών στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να προωθήσει το ρόλο των γυναικών στις αναπτυσσόμενες χώρες. Στα διεθνή φόρα, στη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα. Καμιά φορά πραγματικά έχω την αίσθηση ότι ζω παρεστήσεις με αυτά που ακούω. Ο καιρός είναι πια η ισότητα των φίλων να βρίσκονται στο επίκεντρο της επεξεργασίας των αναπτυξιακών πολιτικών, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών. Ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό η συνάδελφος Ουλσκοκ. Ευχαριστώ. Η έκθεση αυτή δείχνει το πώς οι άντρες και οι γυναίκες προκαλούν με διαφορετικό τρόπο την κλιματική αλλαγή και πως έχουμε διαφορετικές ε, προσβάσεις στις πρώτες ύλες. Πρέπει να τα ερευνήσουμε αυτά τα πράγματα, εάν είναι να αλλάξει η συμπεριφορά μας και ο κόσμος. Αυτό θέλουμε οι περισσότεροι εδώ μέσα. Ακόμα και αν δεν ακολουθούμε την ίδια γραμμή. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλα μέρη στον κόσμο χρειαζόμαστε τέτοια γνώση Έχουμε εμπορικέ και περιβαλλοντικέ συμφωνίες ε, με άλλα μέρη του κόσμου και χρειάζονται και πτυχέ ισότητας. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Κίλ Νίλσεν για την έκθεση αυτή της κλιματικής πολιτικής που είναι κάπως διαφορετική και αυτό είναι καλό γιατί οι πολιτικές λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές εάν ε, γνωρίζουμε τις πτυχές ε, του φύλου. Εάν θέλουμε οι πολιτικές, οι κλιματικές που αποφασίζουμε εδώ πέρα να είναι κάτι παραπάνω από κενά λόγια, χρειαζόμαστε εκθέσεις ε, που θα μας καθοδηγούν στην κατάλληλη κατεύθυνση. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ κύριος Τζανόνι. Ο αγώνας ε, κατά των κλιματικών αλλαγών είναι απαραίτητος ε, για την επιβίωση της γης και η Ευρώπη και όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στρατευτούν για να σταματήσουν την αύξηση της θερμοκρασίας κατά δύο βαθμούς. Αυτό είναι ο μόνος τρόπος ε, για να μειώσουμε τις θεομηνίες, τα μετανεσταυτικά κύματα και όλες τις άλλες καταστροφές που επακολουθούν. Το 70% του φτωχο, των φτωχοτέρων της Ευρώπης είναι οι γυναίκες που στον τρίτο κόσμο παίζουν σημαντικό ρόλο για τη διαχείριση του νερού και στην, ε, για τις οικιακές εργασίες και στη γεωργία. Και οι γυναίκες είναι αυτές που σήμερα πρέπει να δουλεύουν παραπάνω λόγω της ξηρασίας και της έλλειψης νερού. Αυτή η προπτική των φύλων θα πρέπει να ενταχθεί σε όλες τις ε, ε, φάσεις ε, και διαδικασίες ε, του ΟΗΕ κατά την μελέτη των κλιματικών αλλαγών. Κυρία Κλάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Το κλίμα αλλάζει. Οι γυναίκες επηρεάζονται και μπορούν να κάνουν κάτι. Και η συζήτηση γίνεται φεδρή μόνο όταν ακούμε λόγους σαν του κυρίου Γκρίφιν. Η, η έκθεση αυτή είναι σημαντική και το ξέρουμε. Ε, πρέπει να αναζητήσουμε αιτίε και λύσεις. Και βεβαίω οι γνώμες διαφέρουν. Παρά όλες τις διαφορετικές ερμηνείες, ένα είναι σίγουρο. Εάν συνεχίσουμε να καταναλώνουμε τόσες πρώτες ύλε, ε, σύντομα αυτές θα εξαντληθούν. Οπότε ούτως ή άλλως πρέπει να υπάρξει εξοικονόμηση ενέργειας. Ε, η κλιματική αλλαγή δεν επηρεάζει μόνο το περιβάλλον μας. Θα έχουμε επιπτώσεις ε, και κοινωνικές ε, και στον ε, τροφίμο. Θα πρέπει λοιπόν να συμπεριληφθούν περισσότερο γυναίκες εδώ πέρα γιατί οι γυναίκες είναι η μισή ανθρωπότητα. 70% των φτωχότερων και 80% των προσφύγων είναι γυναίκες. Γεγονός είναι πως οι γυναίκες ε, μπορούν να εμπλακούν στην ε, καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής. Επίσης, στον ιδιωτικό τομέα εφαρμόζουν οι γυναίκες τα πράγματα στη βάση, αποφασίζουν ε, πως και τι μαγειρεύεται. Αν σκεφτείτε πως η μισή ενέργεια στις κατοικίες σπαταλιέται, βλέπουμε την σημασία εξοικονόμησης εδώ πέρα. Επίσης οι γυναίκες παίζουν βασικό ρόλο στην ανατροφή των παιδιών. Οι εμπειρίες τους πρέπει να χρησιμοποιηθούν και σε ηγετικέ θέσεις. Αν θέλουμε να βελτιώσουμε τον κόσμο, αυτό γίνεται μόνο με τις γυναίκες. Έχουμε λοιπόν σημαντικές συνδέσεις που γίνονται εδώ πέρα. Και πρέπει να επικεντρωθούμε στο βασικό θέμα. Γυναίκες και κλιματική αλλαγή και όχι ό,τι να είναι εδώ μέσα όπως παραδείγματο χάρη ζητήματα αναπαραγωγής ή ποσοστώσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Μπλίνκεβιτσιούτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Πράγματι δεν συνειδητοποιούμε την πτυχή του φίλου στην καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής. Ο κύριος Γκρίφιν δεν καταλαβαίνει την ουσία του θέματος. Πρέπει εδώ πέρα να εργαστούμε σκληρότερα γιατί βεβαίως δεν έχει συμβεί ακόμα η ενσωμάτωση της διάστασης του φίλου στην πολιτική της ε, κλιματικής αλλαγής. Οι φυσικές καταστροφές μας δείχνουν πως κυρίως ε, τα γυναικόπαιδα πλήττονται από ε, φυσικές καταστροφές και κυρίως στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Οι γυναίκες απασχολούνται στη γεωργία και δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά. Και μετά δεν έχουν ε, επαρκή πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Θα μπορούσαμε λοιπόν να έχουμε δεδομένα που θα μπορούσαν να μας επιτρέψουν να αξιολογήσουμε τις πτυχές του, του φύλου στην κλιματική αλλαγή που πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα της πολιτικής ένωσης. Ε, κυρία Ματέρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η συνέστηση των δεσμών μεταξύ Προβληματική των φύλων και κλιματικών αλλαγών είναι καινούρια και αυτό, γι' αυτό δεν έχει επιφέρει αλλαγές στις κλιματικές πολιτικές. Η διεθνής κατάσταση σήμερα δεν είναι καλή και ο κίνδυνος να μην καταλήξουμε σε διεθνείς συμφωνίες για τις κλιματικές αλλαγές είναι μεγάλος. Εμείς περιμένουμε την διάσκεψη το Ιούνιο στο Ρίο και θεωρούμε ότι η αντίληψη του φύλου θα μπορέσει να συνεισφέρει στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα αποτελέσματα των, της ανισότητας και να καταπολεμήσουμε τις αιτίες τους. Θα πρέπει να έχουμε τα στοιχεία τα στατιστικά στοιχεία για τις γυναίκες για να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε ποιες είναι οι ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους πρέπει να παρέμβουμε, σε ποιες περιοχές, όπως επίσης να δούμε πώς μπορούμε να ορίσουμε την κατανάλωση νερού, για παράδειγμα, ανά οικογένεια. Χρειάζεται βοήθεια και ανάθεση ευθυνών που θα πρέπει να ολοκληρωθούν στις κοινοτικέ πολιτικές, να ενσωματωθούν στις κοινοτικέ πολιτικές. Εγώ εύχομαι ο δεσμός μεταξύ φύλου και κλίματος να ενταχθεί αποτελεσματικά στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο στις πολιτικές, με μεμονωμένες πολιτικές, διότι αυτό καλύπτει όλες τις σφαίρες της ανθρώπινης δραστηριότητας και θα πρέπει να ενταχθεί οριζόντια σε όλα τα σχέδια και τις οικονομικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Παπαδοπούλου, για ένα λεπτό. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, η αλλαγή του κλίματος προκαλεί περιβαλλοντικές και ανθρωπιστικές κρίσεις. Έχει δραματικές επιπτώσεις στι φτωχές χώρε και στους φτωχούς πληθυσμούς. Αναφερόμαστε εδώ ειδικά για τις γυναίκες γιατί αυτές συνιστούν το 85% των θυμάτων από φυσικές καταστροφές λόγω κλιματικών συνθηκών και το 75% των περιβαλλοντικών προσφύγων αντίστοιχα. Στην έκθεση υπάρχουν πολλές και σωστές εισηγήσεις με τις οποίες συμφωνώ όπω παραδείγματο χάρη η πρόταξη για να επικρατήσει μια κλιματική δικαιοσύνη και ένα δείκτης φιλικό προς το περιβάλλον εκείνο το οποίο όμω πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα είναι η ανάγκη να ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου σε όλες τι πολιτικέ για το κλίμα και τη βιώσιμη ανάπτυξη προ τούτο χρειάζονται εξειδικευμένε έρευνε και εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα φύλου για να χαραχθούν ορθολογιστικέ στρατηγικέ πρόληψη και διαχείριση κινδύνων από φυσικέ καταστροφέ για να γίνει σωστή διαχείριση τη περιβαλλοντική μετανάστευση και για να υπάρχει επαρκή χρηματοδότηση από ταμεία και μέσα που συνδέονται άμεσα με το κλίμα η άποψή μου είναι πω η ευρωπαϊκή ένωση πρέπει να ενσωματώσει τη διάσταση του φύλου σε στοχευμένε πολιτικέ για το κλίμα ώστε να δοθούν λύσει. Κυρία Ζαμπόρσκα τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ την εισηγήτρια για τη δουλειά της. Ιδιαίτερα όταν διαβάζω το σημείο 30 Βλέπω ότι λέει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζει ότι η αύξηση του πληθυσμού επηρεάζει και το κλίμα και τονίζει έτσι την ανάγκη να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των γυναικών και ως προς την αντισύλληψη. Εδώ θέλω να αναρωτηθώ, εννοεί η εισηγήτρια ότι πρέπει να πάψει η αναπαραγωγή για να αντιμετωπιστούν οι κλιματικές αλλαγές και να συνδυαστεί η διανομή αντισυλληπτικών με τη μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακος. Η έκθεση αυτή λέει ότι πρέπει οι γυναίκες τελικά να μειώσουν τη θηλυκότητά τους, να μην γίνονται μητέρες, ενώ κανένας από τους στόχους της χιλιετίας δεν λέει ότι πρέπει να μειωθεί η γεννητικότητα η ζωή ενός ανθρώπου έχει την ίδια αξία παντού, ακόμη και αν είναι μακριά από μας ορισμένη. Ε, μπορεί να υπάρχει έλλειψη νερού και άλλα προβλήματα. Πληρώνονται εκατομμύρια για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα, αλλά μία από τις κύριες πηγές της ανέχειας σύμφωνα με τη συντάκτρια και των κλιματικών αλλαγών είναι λέει η αύξηση του πληθυσμού. Αυτό δεν ισχύει και τόσο πολύ γιατί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δημοσίευσε πέρυσι στοιχεία για τις 10 ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες του κόσμου και 7 από αυτές έχουν υψηλή γεννητικότητα. Είναι κρίμα που αυτό υπονομεύει όλα τα υπόλοιπα θετικά στοιχεία της έκθεσης. Ευχαριστούμε. Κυρία Ματζόνη. Ευχαριστώ. Με την έκθεση Κιλ Νίλσεν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδεικνύει για μια ακόμη φορά πόσο αποφασισμένο είναι να υποστηρίξει στη δημιουργία μιας ε, πιο δίκαιης, ε, πιο δημοκρατικής, πιο συμμετοχικής κοινωνίας δεν πρόκειται για ψύχωση όπως είπε ο συνάδελφος Έλμερ, πρόκειται για αποφασιστικότητα να δημιουργηθεί δηλαδή μια Ευρωπαϊκή Ένωση πιο προσαρμοσμένη στις προκλήσεις της τρίτης χιλιετίας. Η έκθεση Νίλσεν στοχεύει στον συνδυασμό του του ζητήματος του φίλου με τις κλιματικές αλλαγές. Εγώ βέβαια δεν κατάλαβα καλά παρά την προσπάθεια της εισηγήτριας αυτούς τους άμεσους δεσμούς. Σημερίζομαι όμως απόλυτα τους ευρύτερους στόχους αυτής της έκθεσης. Δηλαδή να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μία κοινωνία στην οποία δεν θα γίνονται δεκτές οι ανισότητες δεν μπορούμε εμείς να δεχόμαστε μία κοινωνία όπου οι γυναίκες κατέχουν λιγότερο από το 1% των παγκοσμίων αγαθών, όπου πληρώνονται με λιγότερο από ένα δολάριο, όπου είναι μια ελάχιστη μειοψηφία στη θεσμική εκπροσώπηση. Παράγουν όμως το μεγαλύτερο παγκόσμιο εισόδημα εργαζόμενες ε, περισσότερο. Εγώ θεωρώ ότι η έκθεση Νίλσεν αποτελεί καταγγελία όλων αυτών των αδικιών και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μοχλός για να ενεργοποιήσουμε όλα αυτά τα μέσα που ανέφερε ο Επίτροπος Ποτότσνικ για να τα, ε, και να τα εντάξουμε ενεργά σε όλες τις πολιτικές. Διότι το γυναικείο ζήτημα θα πρέπει να λειτουργήσει και να, το, να επαναπροταθεί εγκαρσίως σε όλες τις κοινοτικές προτάσεις και σε όλες τις εθνικές πολιτικές. Η κυρία Πιετικάινεν, την οποία όμως δεν τη βλέπω. Πάμε στο Κατσδιάι. Η κυρία Ρωμάνα Γιορτανσίζο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να πω πως συμφωνώ πως υπάρχει μία σχέση μεταξύ γυναικών και κλιματικής αλλαγής. Συμφωνώ όμως με την κυρία Κρίστα Κλάς. Δεν μπορεί να μείνουμε στις λεπτομέρειες. Πρέπει να δούμε τα σημαντικά ζητήματα. Η εκπαίδευση έχει μεγάλη σημασία λοιπόν ε, λένε πως αν εκπαιδεύσει έναν άντρα έχεις έναν εκπαιδευμένο άνθρωπο και αν εκπαιδεύσει μια γυναίκα έχει μια εκπαιδευμένη γυναίκα. Οπότε έχει σημασία η εκπαίδευση. Η ενημέρωση επίσης είναι σημαντική γιατί έτσι θα επηρεαστούν τα πρότυπα εντός της οικογένειας. Επίσης οι γυναίκες είναι σε μεγαλύτερο βαθμό θύματα της κλιματικής αλλαγής και πρέπει βεβαίως να το προσέξουμε αυτό, ειδικά το μιλάμε για την αναπτυξιακή βοήθεια που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, ε, θα ήθελα να αναφέρω την εκπροσώπηση των γυναικών στη λήψη αποφάσεων. Στηρίζω όλες τις προσπάθειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υψηλότερη συμμετοχή των γυναικών στη λήψη αποφάσεων γενικώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Γεννάκη. Mike, please. Με μικρόφωνο παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Αν μου επιτρέπετε θα ήθελα να αναφέρω κάποια ε, να κάνω κάποιες επικριτικές παρατηρήσεις. Όταν μιλάμε για το κλίμα, συχνά μιλάμε μόνο για αριθμούς και αγορές. Όταν μιλάμε για την κλιματική αλλαγή πρέπει να εστιάσουμε στους ανθρώπους. Οι γυναίκες από τις όμενες χώρες ε, που έχουν, είναι ισχυρότερη θέση και αυτό δεν σχετίζεται μόνο με την αποτυχία των αγορών. Το θέμα είναι το πώς επηρεάζει τις καθημερινές ζωές μας. Και αυτό συχνά το ξεχνάμε. Όταν μιλάμε για κλιματική αλλαγή, μιλάμε για ανθρώπους και μετά είναι οι αγορές και οι αριθμοί. Σας ευχαριστώ. Ρωμέβα. Λοιπόν, καθαρά και εξάστερα. Δεν είναι τυχαίο ότι τα περισσότερα θύματα των θεομηνιών είναι γυναίκες. Αυτό έχει να κάνει με το πόσο ε, είναι αδύναμες οι γυναίκες. Εδώ πρόκειται για τη διαρθρωτική πατριαρχική δομή των κοινωνιών. Ακούσαμε εδώ τοποθετήσεις, οι προτάσεις της κυρίας Νίλσεν είναι βασικές, είναι κοινοτυπίες, είναι διαπιστώσεις. Απαιτούν οι γυναίκες να συμμετέχουν σε όλα τα επίπεδα και αντί να είναι θύματα να γίνουν πρωταγωνιστές να μπορέσουν να επενδύσουμε περισσότερο σε κατάρτιση, προστασία, προετοιμασία και τρίτο να εντάξουμε τις προπτικές του φίλου στον αγώνα ε, για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Πρόκειται λοιπόν για κοινό νου. Και μερικά που μας είπαν εδώ οι συνάδελφοι είναι άλλου αιώνα πράγματα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συγχαρητήρια στην ε, συνάδελφο Κιλ Νίλσεν για αυτήν την εξαιρετική έκθεση. Οι γυναίκες, όπως είπε και η συγγήτρια, πλήττονται ιδιαίτερα από τις κλιματικές αλλαγές. Και αυτό γιατί δεν έχουμε παρκή μέσα στον ε, ε, στις περιβαλλοντικές πολιτικές δεν έχουμε και πολιτικά μέσα δεν έχουμε ε, ανάληψη ευθυνών στον κόσμο και στην Ευρώπη. Να σας πω και κάτι πιο συγκεκριμένο παράδειγμα. Οι γυναίκες στην Αγία, στη χώρα μου, είναι γυναίκες που ψαρεύουν. Και ξέρουμε ότι οι κλιματικές αλλαγές ε, ε, έχει επιπτώσεις και στην κυβερνητική η πολιτική. Η κυβέρνηση δεν πληρώνει, οι γυναίκες αυτές δεν μπορούν να ψαρέψουν γιατί οι ακτές δεν είναι καθαρές. Οπότε υπόκεινται άμεσα τις κλιματικές αλλαγές. Πρέπει να κάνουμε κάτι για να τις βοηθήσουμε. Τελειώσαμε με τη συζήτηση. Να ακούσουμε και πάλι την Κομισιόν. Ο κύριος Ποτόσνικ έχει το λόγο. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα να πω ότι μιλάμε για τις γυναίκες και το κλίμα. Μιλάμε για πραγματικό και σοβαρό πρόβλημα. Γι' αυτό εκτιμώ την προσοχή που έδειξε η συγγήτρια και όλοι εσείς και είμαι σίγουρος πως και η κυρία Χέντεγκάρντε το εκτιμά. Υπάρχουν πολλά πιστικά στοιχεία Αυτά τα οποία μου έμειναν μετά από αυτή τη συζήτηση ήταν κάποιες λέξεις, όπως ενημέρωση, δεδομένα, γνώση, εκπαίδευση, ενσωμάτωση, επιστήμη. Για την στήριξη των γυναικών και της εκπαίδευση των γυναικών μπορώ να προσθέσω πως μέχρι το 2015 θα έχουμε περισσότερες, ε, περισσότερους δείκτες ε, αναφύλλω και ορίζοντας 2020 ε, για τα έργα μας τα κλιματικά θα συμπεριλαμβάνει ανάλυση ένα φύλλο. Κάποιοι από εσά θα γνωρίζετε πως ε, στην προηγούμενη θητεία μου ήμουν υπεύθυνο για την έρευνα και την ε, επιστήμη. Και το ζήτημα των γυναικών στην επιστήμη ήταν πάρα πολύ σοβαρό και προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε. Δυστυχώς δεν υπάρχει εύκολη λύση. Υπάρχουν κάποιες εξελίξεις που είναι πολύ ενθαρρυντικές τώρα. Υπάρχουν κάποια γεγονότα ο αριθμός των ε, γυναικών με διδακτορικά αυξάνεται γρηγορότερα από ό,τι για τους άντρες. Οι γυναίκες ε, ερευνήτριες αυξάνονται με ρυθμό διπλάσιο των ανδρών. Οπότε η κατάσταση βελτιώνεται. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας και στο μέλλον. Αλλά το πρόβλημα βεβαίω ε, αλλάζει όταν περνάνε από τις σπουδές στον κόσμο της εργασίας οι γυναίκες κερδίζουν λιγότερα από τους άντρες να έχουν ε, συμβόλαια μικρότερης ε, διάρκειας, ε, εξελίσσονται αργότερα κτλ. κτλ. Αυτά είναι πραγματικά ζητήματα και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Είναι στην ουσία των πραγμάτων. Και μέσω της κοινωνικής πολιτικής πρέπει να τα δούμε αυτά. Στο μέγιστο βαθμό. Εγώ ίδιος έχω ζήσει την δύναμη των γυναικών στις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Και μπορώ να πω εκ πείρας πως είναι γεγονός. Τέλος, αυτό το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι στο πλαίσιο κάποιου πράγματος που συζητήσαμε χθες. Χθες ήμουν στη Δανία. Είχαμε το άτυπο συμβούλιο που είχε αφιερωθεί σε δύο θέματα. Το ένα ήταν το έβδομο πρόγραμμα ε, πλαίσιο για το περιβάλλον και αφορά το επόμενο επεισόδιο της περιβαλλοντικής μας πολιτικής μέσω μακροπρόθεσμα και το ορίο συν 20. Περίπου το ίδιο δηλαδή, αλλά πιο διεθνές. Μπορώ να πω πως η ισορροπία των φύλων ε, τονίστηκε στις συζητήσεις μας. Πρέπει λοιπόν να τα δούμε αυτά τα ζητήματα όχι μόνο στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής αλλά στο πλαίσιο της πράσινης ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. Όπως σωστά επισημάνατε, η συμπερίληψη, η ισότητα είναι απολύτως απαραίτητες για την βιώσιμη ανάπτυξη. Όπως ακριβώς η ανάπτυξη δεν μπορεί να αφορά μόνο την οικονομία, ούτε και η βιωσιμότητα μπορεί να αφορά μόνο την προστασία του περιβάλλοντος. Η ανάπτυξη πρέπει να εστιάζει στους ανθρώπους, να δίνει δικαιώματα, αξιοπρέπεια και η πράσινη ανάπτυξη πρέπει βεβαίως να είναι ισότιμη και να συνεισφέρει στην εξάλληψη της φτώχειας και να στηρίζει το φυσικό περιβάλλον. Επί τη ευκαιρία ο τίτλος της διάσκεψης ε, στο Ρίο, στο οποίο θα πάμε τον Ιούνιο, στο Ρίο Τετζανέιρο, είναι ακριβώς αυτό. Η πράσινη οικονομία στο πλαίσιο της καταπολέμησης της φτώχειας και τα ζητήματα αυτά είναι πάρα πολύ ε, σημαντικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπε. Πριν ε, δώσω το λόγο στην εισηγήτρια θα ήθελα να πω πως ε, η συζήτηση θα ολοκληρωθεί με μια γυναίκα αντιπρόεδρο βεβαίω. Η κυρία Κιλ Νίλσεν. Εγώ το ήξερα ότι μπορούσαμε να βασιστούμε στην κυρία Χίντεγκαρτ και στην Κομισιόν. Ξέραμε ότι μπορούσαμε να βασιστούμε στην Δανική Προεδρία διότι και έλαβε υπόψη της ε, πολλά από αυτά τα οποία προτείναμε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους, άντρες και γυναίκες ε, που είναι παρόντες σήμερα, που συμμετείχαν στη συζήτηση. Αντικατοπτρίζει το πόσο ε, καρποφόρα ήταν η συνεργασία και το που οδηγεί όλη αυτή η συνειδητοποίηση. Ο καθένας μας εδώ συνεισέφερε σε αυτή την έκθεση και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη. Επίσης ξέρω ότι μπορούμε να βασιστούμε και στο Ίδρυμα για την Ισότητα των Φύλων που δημιουργήθηκε στο Βίλνιους το 2011 και θα ήθελε επίσης να αποτίσω φόρο τιμής σε όλες τις γυναίκες ανά τον κόσμο και στις γυναικείες οργανώσεις που εδώ και πάρα πολύ καιρό κατάλαβαν ότι θα έπρεπε να κινητοποιηθούμε για τα κλιματικά ζητήματα, για την προστασία των φυσικών πόρων Θέλω να αναφέρω το κίνημα ΣΥΠΚΟ στην ε, Ινδία. Οι γυναίκες οι οποίες ε, δέθηκαν ε, στα δέντρα για να προστατεύσουν τα δέντρα, τις γυναίκες στη Ρουάντα που διαφύλαξαν 600 ποικιλίε φασολιών, το κίνημα Χακάρι με την πράσινη ζώνη που προστάτευσε εκατομμύρια δέντρα Εκατομμύρια γυναίκες έχουν λάβει συνείδηση, έχουν συνειδητοποιήσει συγγνώμη, το πρόβλημα ανά τον κόσμο και παλεύουν. Τώρα για το θέμα των ποσοστώσεων. Όσον αφορά στην πολιτική μου ομάδα, εμείς είμαστε υπέρ αυτού του εργαλείου, αυτού του μέσου. Μας επέτρεψε να είμαστε και η μόνη πολιτική ομάδα στο Κοινοβούλιο που έχει ισομέρεια φίλων. Χωρίς το μέσω της ποσόστοσης δεν μπορούμε να έχουμε ισότητα, αλλά πρόκειται απλά για ένα εργαλείο, για ένα μέσο. Και να σας αναφέρω αν μου επιτρέπετε τον Άινστάιν που έλεγε ένα πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί παρά μόνο από το ίδιο επίπεδο συνειδητοποίησης που έχει δημιουργήσει γύρω από αυτό. Ευχαριστούμε πολύ κυρία εισηγήτρια. Έληξε η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα στις 12 το μεσημέρι. Και περνάμε στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη, που είναι η